Παρακαλώ καθίστε. Επαναλαμβάνεται η συνεδρίαση που διακόπηκε στις 12 ε, Δεκεμβρίου τα πρακτικά και τα κείμενα που εγκρίθηκαν στις 12 ε, Δεκεμβρίου είναι στην διάθεσή σας. Υπάρχουν αντιρρήσεις. Μου λένε πως δεν υπάρχει διερμηνία στα αγγλικά.